So, και αγαπητοί συνάδελφοι, σα παρακαλώ καθίστε. Θα αρχίσουμε αμέσως την συνεδρίασή μας, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου δηλαδή, με πρώτο θέμα την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Επειδή είναι αυτή η υπερπλήρης και έχουμε και ορισμένα σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε με τους συντονιστές, θα προτείνω να αναβάλουμε το υπαριθμό 5 για να το συζητήσουμε σε κάποιο ιστερότερο χρονικό σημείο. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε. Ψήφι υπέρ της αναβολής του υπαριθμών 5. Σας ευχαριστώ. Σαφής η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αναβάλλεται λοιπόν η συζήτηση του 5. Υπάρχουν άλλα σχόλια για την ημερησία διάταξη. Δεν υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη και έρχομαι στο υπαριθμόν 2, όπως συνήθως. Έγκριση λοιπόν των πρακτικών της συνεδριάσεως θα θεωρήσω ότι έγινε εάν μέχρι τέλους της συνεδριάσεως δεν έχουν εγερθεί ενστάσεις. Ακολουθεί το 3. Υπενθυμίζω ότι μεταδίδεται διαδικτυακώς η συνεδρίασή μας και είναι πιθανόν να σας παρακολουθούν τώρα που εργάζεστε εδώ ένας αριθμός ε, θεατών. Έχω και ορισμένες άλλες σύντομες ανακοινώσεις για την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδιών και για τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Υπάρχει κάποια κίνηση εκεί και αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματευτές συναντήθηκαν ξανά στις 18 πρώτου και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά. Η δε συμφωνία TTIP είναι πλέον ε, κοινού ενδιαφέροντος όσο γνωρίζετε ενδιαφέρονται όλοι και ο επόμενος γύρος θα διεξαχθεί στις 22 του μηνός εδώ στις Βρυξέλλες. Ελπίζω τα ευαίσθητα θέματα τότε να αποτελέσουν επίσης αντικείμενο των σχετικών διαβουλεύσεων. Εδώ ε, οφείλω να σημειώσω μία εξέλιξη που έχει σχέση με την ροή δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Ενωμένων Πολιτειών. Θα θυμάστε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέτρεψε ως μη νόμιμη την ε, συμφωνία του ασφαλούς λιμένος, safe harbor στα αγγλικά. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό όταν θα έχουμε το κείμενο, το τελικό κείμενο. Το ζήτημα του επόμενου γύρου των περιβαλλοντικών αγαθών επίσης έχει προγραμματιστεί για 3 και 4 Μαρτίου ώστε και εδώ θα πρέπει να αναμένονται κάποια βήματα πρόοδου. Η Συμφωνία Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσης Βιετνάμ έχει ήδη δημοσιευτεί και νομίζω ότι μπορεί έτσι κανείς να εξετάσει και τα διάφορα στοιχεία όπως το κεφάλαιο περί αηφορίας. Ακολουθεί το θέμα υπαριθμών 4 έχω την ευχαρίστηση να ευχηθώ το καλώς ορίσατε στην κυρία Πολάσκη, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία βρίσκεται εδώ κοντά μας. Καλώς ορίσατε λοιπόν κυρία Πολάσκη. Έχουμε ορισμένες, έχουμε διεξαγάγει ορισμένες στρατηγικές συνομιλίες για θέματα εμπορικής πολιτικής εδώ στον 21ο αιώνα. Έχουμε υποδεχτεί τον Πασκάλ Λαμί, Μάρι Νίμι, δηλαδή Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ο ΟΣΑ. Και ένα σημαντικό στοιχείο της εμπορικής μας πολιτικής για τον 21ο αιώνα είναι βεβαίως και τα θέματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η διατήρηση και εφαρμογή του, της θεμελιώδους συνθήκης του ILO. Σε αυτά τα θέματα θα έρθουμε τώρα σε ό,τι αφορά τις εμπορικές προτιμήσεις στα πλαίσια του ESP και θα διεξαγάγουμε και μια κοινή ακρόαση. Έτσι λοιπόν ε, το ερώτημα της εφαρμογής των προτύπων ILO έχει μεγάλη σημασία για την διατήρηση της πορείας της εμπορικής μας πολιτικής. Σας ευχαριστώ που είστε παρούσα εδώ και σας παραδίδω το μικρόφωνο. Uh, good afternoon. Uh, let me start by thanking... Καλησπέρα σα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και τον Πρόεδρο, τον κύριο Λάγκε, για την ευκαιρία να σα ευχαριστήσω σήμερα. Νομίζω το πιο χρήσιμο θα ήταν να σα παρουσιάσω μια επισκόπηση του ρόλου του ILO και των θεμάτων εργασία για την παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε και το θέμα είναι να σας πω πώς την ε, συνδυάζουμε και πώς μπορούμε να χρησιμεύσουμε στη δική σας τη δουλειά αυτή της Επιτροπής και άλλων κυβερνήσεων που έχουν να κάνουν με εργασιακά θέματα, κοινωνικά και άλλες ε, σχετικές υποθέσεις. Ε, θα σας κάνω λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις. Ο ΑΕΛΟ δίνει μεγάλη σημασία στην ε, δουλειά της Επιτροπής σας. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου αυτής της Επιτροπής όλο ιδιαίτερος και ημών έχει αναπτυχθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλούς, πολλοί από τους συναδέλφους μου του ΑΕΛΟ ήδη έχουν έρθει εδώ για να συζητήσουν μαζί σας και αύριο θα συζητήσουμε και το θέμα του GSP Plus με παρουσία των μελών της Επιτροπής σας. Ο ΑΕΛΟ λοιπόν θα συνεχίσει να στηρίζει την Επιτροπή σας σε θέματα που έχουν να κάνουν και με, το δικό μας, με τη δική μας εντολή. Όπως ξέρετε, σύντομα θα συμπληρώσουμε τα 100 έτη ηλικίας μας, όπως προέβλεπε η συνθήκη των Βερσαλιών όταν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πεποίθηση του προημίου ε, του συνθετική μα συνθήκη του 1919 έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ανθρώπινε συνθήκε στην εργασία. Ιδάλω ε, θα υπάρχει ε, εμπόδιο για τα οποιαδήποτε άλλα έθνη θέλουν να βελτιώσουν τι εργασιακέ συνθήκε στη χώρα του. Ελπίζω να συμφωνείτε ότι και στην παγκοσμιοποίηση του 21ου αιώνα αυτό ισχύει όπω ίσχυε το 1919. Ε, τώρα, το 1988 185 μέλη είχε πλέον διάθεση του ΑΕΛΟ και πάρα πολλές οργανώσεις και ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Έτσι απηχούμε και τις δημόσιες και τις ιδιωτικές απόψεις και εγκρίναμε μια δήλωση, τη δήλωση για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στον χώρο εργασίας, η οποία καθορίζει τέσσερα βασικά εργασιακά δικαιώματα τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλε τι χώρε. Αυτό συμφωνήθηκε από όλε τι χώρε, ασχέτω του επίπεδου οικονομική ανάπτυξη και του αν είχαν κυρώσει τι βασικέ μα ε, συμβάσει και συνθήκε ή όχι. Αυτό θεωρήθηκε μια βασική συνιστόσα των προσπαθειών να διατηρήσουμε τον συνδυασμό μεταξύ κοινωνική προόδου ε, οικονομική ανάπτυξη και τη ε, προϊούσα παγκοσμιοποίηση η ελευθερία του συνασπίζεστε, η πραγματική αναγνώριση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η εξάλληψη τη υποχρεωτική ή καταναγκαστική εργασία, η κατάργηση τη παιδική εργασία και η κατάργηση τη διακριτική μεταχείρισης ε, στην απασχόληση. Ήταν τα τέσσερα βασικά δικαιώματα που ορίστηκαν από οκτώ εργασιακά πρότυπα, τα οποία ονομάζουμε βασικέ συμβάσει, core συμβάσει. Από τότε όλοι οι συμβαλόμενοι ενέκριναν δηλώσεις για την κοινωνική δικαιοσύνη στα πλαίσια μιας ε, δίκαιας παγκοσμιοποίησης. Αυτό που ονομάζεται και αξιοπρεπής εργασία. Η αξιοπρεπή εργασία συμπεριλαμβάνει το σεβασμό για αυτά τα βασικά εργασιακά δικαιώματα που μόλι ανέφερα, αλλά επίση συμπεριλαμβάνει την προώθηση των δυνατοτήτων απασχόληση, την κάλυψη τη κοινωνική προστασία για όλου του ε, ανθρώπου και τον κοινωνικό διάλογο καθώ και την ε, ισότητα στον χώρο εργασία. Αυτή η αρχή διέπει την εργασία όλων των μελών του ΑΕΛΟ και των μελών του Προεδρείου μα την κατάρτιση των ε, οικονομικών του πολιτικών και των εμπορικών του πολιτικών ω προ τον αντίκτυπο που έχουν στι εργασιακέ συνθήκε και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η δήλωση αυτή ε, προσφέρει τη δυνατότητα στον ILO να μπορέσει να συνδράμει τα μέλη που θέλουν να βελτιώσουν τα εργασιακά του στα πλαίσια πολυμερών ή διμερών ε, εμπορικών συμφωνιών, άλλων εμπορικών συμφωνιών και πάντοτε ανάλογα με το κατά πόσο όλα αυτά είναι συμβατά με την εντολή και τι υποχρεώσει του ΑΕΛΟ. Με, αυτή τη συγκεκριμένη εντολή έχουμε πραγματοποιήσει συγκεκριμένε έρευνε για τα εργασιακά θέματα τα τελευταία χρόνια, πολλέ φορέ και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον ΠΟΕ, και με άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Ε, οι έρευνες αυτές δείχνουν διαρκώς ότι πρέπει να επιδιώκουμε την εμπορική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη πάντοτε ε, σε έναν συνδυασμό με, τα με τις κοινωνικές μας μέρημνες. Οι συνεπείς κοινωνικές ε, πολιτικές μπορούν να κάνουν την εμπορική πολιτική πιο ανοιχτή και να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, σεβασμό των εξωτερικών δικαιωμάτων, μεγαλύτερη ισότητα και μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο. Ενώ μπορεί να προκύπτουν και οικονομικέ ευκαιρίε για τι χώρε και τι εταιρείε. Για να επιτέχουμε του στόχου αυτού, υπάρχουν, υπάρχουν εργασιακέ ρήτρε σε πολλέ πολυμερεί, περιφερειακέ και διμερεί εμπορικέ συμφωνίε τα τελευταία χρόνια, όπω τα γνωρίζετε. Ε, ήδη από το 2013, πάνω από το 80% όλων των εμπορικών συμφωνιών που τίθενται σε ισχύ συμπεριλαμβάνουν εργασιακέ και ε, κοινωνικέ ρήτρε και απαιτήσει. Αυτή η ανάπτυξη εν μέρει οφείλεται στο γεγονό ότι πολλέ εμπορικέ συμφωνίε έχουν ε, αποτελέσει αντικείμενα διαπραγμάτευση μεταξύ των χωρών που ε, προσχωρούν σε αυτέ τι κοινωνικέ ρήτρε, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα και ο Καναδά, αλλά και άλλε αναπτυσσόμενων οικονομιών όπω ε, οι που επιλέγουν να συμπεριλάβουν τέτοιες ρήτρες, ακόμη και στις δικές τους συμφωνίες μεταξύ τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένα εργαλεία του ILO, συγκεκριμένα τη δήλωση του 1988 που ορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της εργασίας, αλλά και την δήλωση του 2008 που καθορίζει την αρχή της αξιοπρεπούς εργασίας με πολλές εμπορικές συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτά τα βασικά εργαλεία και πρότυπα αλλά και συμβάσεις προκύπτει μια σημαντική ευκαιρία για να υπάρχει συνοχή και σύγκληση σε όλο το φάσμα εμπορικών συμφωνιών που μπορεί να συνάπτονται σε όλες τις διαφορετικές χώρες. Όμω προκύπτουν και προβλήματα ω προ την υλοποίηση και την εφαρμογή των ρητρών αυτών με τρόπο εύρωστο και συνεπή σε όλο τον πλανήτη και που να είναι και συνεπή με τι ανάλογε συμβάσει του ΆΕΛΟΥ. Υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ΆΕΛΟΥ έχει ε, και ένα σύστημα ε, παρακολούθηση επίβλεψης για να αντιμετωπίσει τις προσφυγές των κρατών μελών που δεν έχουν σεβαστεί τις ε, συμβάσεις που κύρωσαν ή τα πρότυπα εργασία που έχουν προβλεφθεί. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε εργαζόμενο, από οποιαδήποτε ήπειρο, με διαφορετικά νομικά συστήματα ή με διαφορετική προσέγγιση στα εργασιακά δικαιώματα στον εργασιακό χώρο. Υπάρχει λοιπόν μια βασική εμπειρογνωμοσύνη που ε, προσφέρεται για το κατά πόσο υπάρχει συμβατότητα με τα διεθνή εργασιακά πρότυπα ή τη μη συμμόρφωση και τι ε, εικόνα μπορεί να παρουσιάζει αυτή στην πραγματικότητα. Πέραν αυτών των αναφορών στα βασικά εργασιακά δικαιώματα και την αρχή τη εξωτερική εργασία, πολλέ εμπορικέ συμφωνίε περιλαμβάνουν και διατάξει που έχουν να κάνουν με το διάλογο και την τεχνική αρρωγή, προκειμένου να ενδυναμωθούν τα εργασιακά δικαιώματα, ιδίω σε χώρε που είναι εμπορικοί εταίροι. Αυτέ οι ρήτρε κάποιε φορέ ε, συμπεριλαμβάνουν και την συμμετοχή του ILO. Πολλέ φορέ όταν αναφέρεται σε μια συμφωνία ο ILO, αλλά και όχι, ε, ήδη η παρουσία του είναι αισθητή. Είμαστε παρόντε σε πολλέ χώρε ε, μέλη μα, ιδίω τι αναπτυσσόμενε, που χρειάζεται να ενισχύσουν την νομική προστασία των δικαιωμάτων και την πρακτική εφαρμογή υλοποίηση αυτών. Οπότε όταν οι εμπορικοί εταίροι έρχονται σε εμά και μα ζητούν τη βοήθειά μα, πολλέ φορέ δεν χρειάζεται να πάνε και πολύ μακριά. Θα βρουν ένα γραφείο του ΑΕΛΟ στη χώρα του και κάποιον πρόσωπο του ΑΕΛΟ που είναι πολύ κοντά του και γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν επί στη χώρα ή τι τεχνικέ δυσκολίε μπορεί να παρουσιάζονται και να προτείνει και λύσει. Μπορεί να κοιτάξουμε να δούμε τώρα περισσότερο λεπτομερό την συνεργασία ΕΛΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι πολλέ οι χώρε που, όπω είπα, ε, συμπεριλαμβάνουν τι ρήτρε του ΑΕΛΟ και ζητούν τη συνεργασία του ΑΕΛΟ. Ο ΑΕΛΟ καλωσορίζει την συμπερίληψη σε πολλέ εμπορικέ συμφωνίε και προτιμησιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζει τι μνήμε και την αναφορά στα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Προκειμένου αυτά να υλοποιούνται στην εθνική νομοθεσία με τρόπο συνεπή κατά τα διεθνή εργασιακά πρότυπα. Ένα παράδειγμα ένα καλό παράδειγμα συνεργασία σε τέτοιε πολιτικέ ε, από Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα αιτήματα που έχουν αποφυνθεί στον ΑΕΛΟ για την Κορέα, η FTA τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Κορέα ή το αίτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη προ του εταίρου γύρω από το θέμα τη διακριτική μεταχείριση για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν όταν χρησιμοποιήθηκε η σύμβαση του ΑΕΛΟ 111 κατά τη διακριτική μεταχείριση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συνεργασία μεταξύ του ΑΕΛΟ και της ε, DG Trade, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, με το σύστημα των ενισχυμένων προτιμησιακών, της ενισχυμένης του ενισχυμένου προτιμησιακού συστήματος. Εδώ ε, η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων καθώς και των, βασικών, των οκτώ βασικών συμβάσεων του ΑΕΛΟ είναι ένα αντικείμενο που μας απασχολεί και στη συνεργασία μας με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου κοιτάζουμε οι χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα αυτό, το Γουατεμάλα, το Πακιστάν, η Μογγολία και η Νότια Κορέα να δούμε κατά πόσο οι τέσσερι αυτέ χώρε ε, συμμορφώνονται με τι υποχρεώσει του των ε, βασικών συμβάσεων σύντομα θα καλύψουμε και την Αρμενία, τις Φιλιππίνες, το, το πράσινο κροτήρι και την Παραγουάη. Εδώ ο ΑΕΛΟ καθορίζει μια νέα εμπορική στρατηγική που θα δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο ε, με την φιλοδοξία να υπάρχει καλύτερη συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα και την ε, ε, καταγραφή αυτών σε διεθνές επίπεδο με όλες τις χώρες εταίρους, καθώς και αυτά να μεταφραστούν στην έννοια της εξωπροπούς εργασίας, με τα βασικά εργασιακά δικαιώματα και τον κοινωνικό διάλογο και τις ευκαιρίες και την κοινωνική προστασία επιπλέον. Επίσης, καλωσορίζουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις υπεύθυνες ε, αλυσίδες προμήθειας, όπως έχουν ονομαστεί. Και να στραφώ λίγο σύντομα στο θέμα αυτό. Ε, το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπορικές σχέσεις 3.000 ετών μεταξύ υπήρων και διαφορετικών περιοχών του κόσμου. Όμως ε, το σύστημα της παγκοσμιοποίησης έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν καθορίζουμε τις εργασιακές ρήτρε και τα εργασιακά δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα το τέλος του ψυχρού πολέμου και η εξέλιξη των οικονομικών πολιτικών στην Κίνα έχουν αλλάξει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού που ήταν διαθέσιμο για να συμμετάσχει στις οικονομίες της αγοράς. Οι εκτιμήσεις λένε ότι οι εταιρείε διαθέτουν το διπλάσιο ή τριπλάσιο εργατικό δυναμικό και τετραπλάσιο σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Πρόκειται για ένα σοκ λοιπόν στο σύστημα από την προσφορά εργατικού δυναμικού, κάτι που άρχισε να ισχύει από τον 21ο αιώνα κατά κύριο λόγο. Οπότε όλοι οι βασικοί νόμοι της αγοράς έχουν μια τεράστια αλλαγή στην ζήτηση, ε, στην προσφορά μάλλον, αλλά αν δεν υπάρχει ανάλογη ε, ανάπτυξη της ζήτηση, και αυτό υπήρχε για κάθε τομέα της οικονομίας, θα υπάρχει μεγάλη πίεση προς τους μισθούς. Τέτοιο σοκ λοιπόν έχουν δεχτεί χώρε όπου το βιωτικό επίπεδο, οι μισθοί ε, όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομίας ήταν πολύ χαμηλότερα, ήταν δηλαδή αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις χώρες που είχαν ήδη υψηλό βιωτικό επίπεδο. Ξέρετε ότι με τις τεχνολογίες πληροφορίας επίσης και τις δυνατότητες ε, ταξιδίων και μετακίνησης που υπάρχουν πλέον, οι εταιρείε έχουν δημιουργήσει συστήματα που είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και μπορεί να απασχολούν εκατοντάδε ω χιλιάδε εταιρείε προμήθεια που να συνεργάζονται μεταξύ του παντού ε, στον πλανήτη. Ω προ τον εργασιακό χώρο, δεν έχουμε ε, βασικά δεδομένα για το οι άνθρωποι μπορούν να συνεργάζονται σε τέτοιε αλυσίδε όπω ονομάστηκαν ε, σε διεθνέ επίπεδο. Όμω έχουμε τουλάχιστον 40 χώρε με βασικά στατιστικά στοιχεία που μα επέτρεψε να απεμπλέξουμε την όλη κατανομή των αλυσίδων αυτών σε πλανητικό επίπεδο για να δούμε πώ διαμορφώνονται οι εγχώριε αλυσίδε σε κάθε χώρα. Περίπου 40 είναι λοιπόν χώρε που απασχολούν 40 εκατομμύρια ανθρώπου ε, σε όλο τον πλανήτη. Μάλλον έχουμε φτάσει στα 300 εκατομμύρια τώρα πια σε σχέση με 140 εκατομμύρια στο παρελθόν. Αυτό συμπεριλαμβάνει πλέον και τι αναδυόμενε οικονομίε και ένα μεγάλο μερίδιο αυτή τη προσφορά εργατικού δυναμικού είναι γυναίκε. 40% περίπου όλων των εργαζομένων σε αυτέ τι 40 χώρε κατά μέσο όρο είναι γυναίκε. Αυτή η παγκοσμιοποίηση του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής έχει δημιουργήσει νέα ανοίγματα οικονομικής ανάπτυξη και έχει αλλάξει και το πρότυπο της εργοδοσίας αλλά και της καταπολέμησης της φτώχειας για εκατομμύρια ανθρώπους. Ταυτόχρονα ελό εκτιμά ότι περίπου 785 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες που εργάζονται σε πλήρη χρόνο δεν έχουν αρκετό χρόνο για να βγάλουν τα νοικοκυριά τους, τα σπίτια τους τι οικογένειέ του από τη φτώχεια δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν κάποια προβλήματα να παραμένουν και να πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πολλοί άνθρωποι αυτοί ε, που ε, ζουν σε συνθήκε φτώχεια εργάζονται σε αυτέ τι παγκόσμιες αλυσίδε προμήθεια. Και ενώ έχουν εξαπλωθεί αυτέ οι αλυσίδε και υπάρχουν εργασιακέ ευκαιρίε, υπάρχουν και ανταγωνιστικέ πιέσει που καταπιέζουν τις τιμές ε, που πληρώνουν οι παραγωγοί και αυτό βεβαίω έχει να κάνει και με του μισθού που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Έτσι, οι εταιρείε προμήθειας αγνοούν τους, τα εργασιακά πρότυπα ε, προσλαμβάνουν σε συνθήκε ανασφάλεια, του αναγκάζουν να εργάζονται σε ε, ωράρια που του εξαντλούν και δεν σέβονται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπω το δικαίωμα του συνασπίστε, την παιδική εργασία, την καταναγκαστική εργασία. Έτσι υπονομεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά εκτό από αυτού που πλήττονται άμεσα, υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό για του υπόλοιπου που θέλουν ε, να ε, εμπορευτούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να έχουν μαζί μα εμπορικέ σχέσει, αλλά και τι κυβερνήσει που θέλουν να σεβαστούν τα εργασιακά πρότυπα σε σχέση με το εργατικό του δυναμικό. Οι βασικέ εταιρείε που ορίζουν τι ευκαιρίε. Του όρου ε, σε αυτέ τι αλυσίδε παραγωγή λαμβάνουν τι αποφάσει παραγωγή ό,τι αφορά το τι επιθυμούν να πληρώσουν, χρόνους παραδόσεων, που μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ αρνητικές συνέπειες στην άλλη άκρη της ε, αλυσίδας της παραγωγής, χωρίς να είναι ταυτόχρονα άμεσα υπεύθυνε για τις επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών. Γνωρίζουμε τις μεγάλες ετικέτες των ε, ε, Αμερικανών και Ευρωπαίων κατασκευαστών ετικέτες, ξαναλέω, που βρέθηκαν στα ερήπια κτηρίων που καταστράφηκαν μετά από σεισμούς ή πυρκαγιές και όπου δούλευαν και παιδιά. Έτσι λοιπόν αυτή η δραματική αύξηση της απασχόλησης οδηγεί και τις χώρες, μάλλον οι χώρες δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική τους αρμοδιότητα. Και σε αναπτυγμένες οικονομίες η μεγάλη ταχύτητα της αλλαγής της αγοράς αυτής μείωσε τις ικανότητες των κρατών να ρυθμίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις συνθήκες όπου εργάζονται. Διαμεθοριακές ε, λοιπόν προσπάθειες και κυβερνήσεων οι οποίες συμμετέχουν σε διεθνείς συμφωνίες έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Ο ILO έχει συλλέξει σημαντική εμπειρία σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα βελτίωση των συνθήκων σε αυτές τις παγκόσμιες συνθήκες παραγωγής. Αυτά που έχουμε διδαχθεί από τις τελευταίες δεκαετίες των εμπειριών μας είναι ότι είναι δυνατόν αυτό, αλλά όχι εύκολο. Έχουμε δει πολλές καλές προθέσεις που δεν οδήγησαν σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Δύο επιτυχημένα παραδείγματα ωστόσο που μας δείχνουν τι, μπορεί, τι, χρειάζεται μάλλον, για να βελτιωθούν οι συνθήκες στις supply chains μέσω συμφωνιών εμπορικού χαρακτήρα. Πρώτο πρόγραμμα μεταξύ του ILO και της International Finance Corporation που γνωρίζετε ότι σε αυτήν συμμετέχει η Παγκόσμια Τράπεζα και που ε, απευθύνεται στους εργαζόμενους στην παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής ρούχου και παπουτσιού με στόχο να γίνει αξιολόγηση των συνθήκων οι οποίοι τις εργάζονται. Έχουμε 1.200 εργοστάσια σε 8 χώρες και περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Αυτοί οι επιθεωρητές αναφέρονται σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση την έκθεση υποβάλλουν και στο εργοστάσιο και στους αγοραστές των προϊόντων δίνουν μια προθεσμία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και μετά κατονομάζουν στις εκθέσεις το εργοστάσιο το οποίο παραβιάζει σοβαρά τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων και αυτά τα αναρτούν στο διαδίκτυο για να τα δει ο καθένας. Διαφάνεια λοιπόν που σημαίνει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής. Είτε πρόκειται για τον παραγωγό, είτε για τον πελάτη, είτε για την κυβέρνηση κάποιας χώρας και ούτω καθεξής. Είναι πολύ αποτελεσματική η προσπάθεια αυτή. Δίνει επίσης το πρόγραμμα δυνατότητα εκπαίδευσης και των μάνατζερ και των εργατών στα εργοστάσια για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις βελτιώσεις. Υπάρχει και τριμερής, ε, δημιουργούνται μάλλον και τριμερής επιτροπές και στο επίπεδο του εργοστασίου αλλά και στο εθνικό επίπεδο της κάθε χώρας με συμμετοχή εκπροσώπων και των εργοδοτών και των εργαζόμενων και είναι το πρώτο βήμα για τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε χώρες όπου δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μπορώ να σας δώσω και παραδείγματα, μπορώ να σας πω και για ορισμένα από τα μετρήσιμα αποτελέσματα στην Καμπότζη για παράδειγμα στα πλαίσια της ε, Συμφωνίας Εμπορίου του 2001 το δεύτερο παράδειγμα που θα μου επιτρέψετε να σα εξηγήσω σύντομα προέρχεται από την κατάρρευση του συγκροτήματος Ράνα Πλάζα πριν από τρία χρόνια στο Μπαγκλαντές που σκότωσε περίπου 1.300 εργαζόμενους και εργαζόμενες. Ε, φάνηκε τότε ποιο είναι το μέγεθος των κινδύνων που κρύβουν οι διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. Ο ILO αμέσως ήλθε σε επαφή με τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων στο Μπαγκλαντές για να συζητήσει τα θέματα και μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριέλαβε και το Global Sustainability Compact το οποίο, στο οποίο συμμετέχουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλοι διεθνείς φορείς για να εξασφαλιστούν δικαιώματα των εργαζόμενων, όπως για δικαιώματα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε, αλλά και για να ληφθούν μέτρα ασφάλειας της υγείας και της ε, σωματικής ακαιρότητας των εργαζόμενων. Μετά από τρία χρόνια από την σύναψη του συμφώνου έγινε μια πρώτη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση βρήκε, ας πω, το μπουκάλι μισογεμάτο, ίσως ούτε καν μισογεμάτο με πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν. Αν έχετε ερωτήσει να μου κάνετε θα σας πω κι άλλα. Ο ILO πρόσφατα ξεκίνησε το Better Work Program, είναι το άλλο παράδειγμα το οποίο ήθελα να σας πω πάλι στο Bangladesh και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα απογεμίσει το μπουκάλι. Τελειώνοντας να σας πω ότι τον Ιούνιο φέτος στην ετήσια παγκόσμια διάσκεψή μας θα συζητήσουμε το θέμα των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής με πάνω από 150 συμμετοχή πάνω από 150 κυβερνήσεων και των δικών σας βεβαίως οργανώσεων ε, εργοδοτών για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε συγκεκριμένα ποιες είναι οι προκλήσεις και ελπίζω μάλιστα να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες συστάσεις που θα μπορούν να εφαρμόζονται για να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις των global supply chains και στην απασχόληση και στην βιωσιμότητα της απασχόλησης. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και αναμένω τις ερωτήσεις σας a real pleasure to listen. Θα δώσω τώρα το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Καταρχήν το ΕΛΚ. Δεν είναι εδώ ο συντονιστής, δεν είναι. Ε, παρόν ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ. Κυρία Πολάσκη, για τις διεξοδικές ε, πληροφορίες. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση για να μου πείτε τη γνώμη του ΔΟΕ σε σχέση με την, ε, το καθεστώς της οικονομίας αγοράς στην Κίνα, κατά πόσο θα της χορηγηθεί αυτό το καθεστώς. Από όσο γνωρίζουμε δεν πληρεί τους όρους για πολλούς ε, λόγους. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε δηλαδή για κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping. Υπάρχουν πολλές ε, χώρες που δεν ε, αποδέχονται αυτό το καθεστώς όπως ο Καναδάς, το ΙΠΑ και μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που πλήττονται και εργαζόμενος, Θα ήθελα να μου πείτε τι γνώμη έχει τη στιγμή που δεν αναγνωρίζετε αυτό το καθεστώς από πολλές χώρες. Ε, David Martin από τους σοσιαλιστές. Ε. Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα σε σχέση με την τήρηση των συμβάσεων του ε, ΔΟΕ από το Ιράν. Στη Γαλλία τα τέλη Ιανουαρίου έγινε ε, λόγος για ένα ε, γαλλικό συνδικάτο που μίλησε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση στο Ιράν, όπου φαίνεται ότι πολλοί συνδικαλιστές αυτή τη στιγμή έχουν φυλακιστεί και θα θέλαμε ε, εδώ ενώπιόν σας να μιλήσουμε για τους ε, βασικούς όρους και συνθήκες που τηρούνται και από πλευράς ΔΟΕ και, στην, ε, και στο Ιράν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλήττονται αυτοί οι συνδικαλιστές και αύριο το πρωί εδώ και από πλευράς ε, η ε, Επιτροπής, ε, συγγνώμη, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι εδώ παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να φυγεί αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να, τήρουν, να τηρούνται αυτά τα δικαιώματά Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα από κοινού. Θα ήθελα να κυρωθεί ακολουθούν οι βασικές ε, συμβάσεις εάν πληρούνται οι όρια. Αυτό ε, χρειάζεται ακόμα να υπάρχει πλήρης κύρωση των συμβάσεων. Όταν μιλάμε λοιπόν για εμπορικές συμφωνίες με αυτές τις ε, χώρες, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών με τις αναπτυσσόμενες χώρες τη στιγμή που πολλές ε, χώρες θεωρούν ότι οι πλούσιες προσπαθούν να επιβάλλουν τους όρους τους και αντί να τους βοηθήσουν ε, προσπαθούν να επιβάλλουν τα δικά τους δεδομένα. Μιλάμε για τη θεωρία της κότας και του αυγού δηλαδή. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές τις χώρες να τηρήσουν αυτές τις προδιαγραφές. Αυτό επιβραδύνει την ε, οικονομική ανάπτυξη. Ελπίζουμε όμως να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, καταρχήν σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Μιλάμε για το εμπόριο το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσει την ευμερία των ανθρώπων υπό την ευρύτερη έννοια και να τηρούμε βασικές αξίες. Πώς βλέπετε το εμπόριο υπό την ευρύτερη έννοια μπορεί να προωθήσει την ευμερία των ανθρώπων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανθρωπιστικές ρήτρες που συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες από όσο γνωρίζετε. Η Αίγυπτος έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις του ΔΟΕ, αλλά δεν τις στηρεί. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος να χάσουμε την αξιοπιστία μας τη στιγμή που προσυπογράφουν οι χώρες, αλλά δεν τηρούν τις συμβάσεις και που υπάρχουν ε, οι υπογραφές επί χάρτου, αλλά επειδή δεν τηρούνται οι συμβάσεις, ε, τότε αποδυναμώνεται το πλαίσιο τη στιγμή που οι χώρες δεν θέλουν να δεχτούν αυτά τα πρότυπα και προδιαγραφές και δεν τα τηρούν. κυρία Μίνα. Μίνα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας, κυρία Πολάσκη. Όπως ξέρετε, ε, αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε πολλές συνθήκες με χώρες, προσχέδια δηλαδή έχουμε συνθήκων, τα οποία βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Για παράδειγμα, τι γίνεται στην περίπτωση της ε, ΤΙΣΑ ε, και της Νότιας Κορέας. Εδώ μιλάμε για το γεγονός ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υπογράψουν τις βασικές συνθήκες και αυτό αφορά και τη Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, την ΤΙΣΑ. Πώς μπορούμε να εργαστούμε. Ζανίκ. Ευχαριστώ. Στην εισήγησή σας μιλήσατε για αξίες και πράγματι Εάν κατά τη δεκαετία του 90 θεωρούσαμε ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου, την απελευθέρωση του εμπορίου και τις συμβάσεις με, τον, με τη ΣΥΠΑ θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μία απελευθέρωση του εμπορίου και αυτό θα οδηγούσε παράλληλα και σε μία πολιτική ε, φιλελευθεροποίηση με στα πλαίσια και των ε, συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ΒΟΕ. Δυστυχώς όμως ε, δεν ε, ίσχυσε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες συμμετέχουν στα πλαίσια των ελευθέρων συναλλαγών και του οικονομικού φιλελευθερισμού, αλλά πρόκειται για ολοκληρωτικά καθεστώτα που δεν δέχονται τις ε, τα προστάγματα του ΔΟΕ. Θα θέλαμε λοιπόν να μιλήσουμε και για τις ελεύθερες συναλλαγές μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θεωρείτε ότι σε αυτή την περίπτωση στις διαπραγματεύσεις, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ή τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ρήτρες για το δικαίωμα στην εργασία. Όταν έγινε μια συζήτηση στο Στρασβούργο, στο Κοινοβούλιο, για την συμφωνία ΤΙΖΑ, για τις συναλλαγές στον τομέα δηλαδή των υπηρεσιών, ο Επίτροπος Εμπορίου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι συμβάσεις του ΔΟΕ. Αυτό όμως δεν μπορεί πλέον να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της Κομισιόν το μας είπε ο Επίτροπος Εμπορίου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΣΑ μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις προδιαγραφές και τις αξίες. Κατά πόσο κρίνεται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό για να τηρηθεί το δικαίωμα στην εργασία παντού στον κόσμο. Ευχαριστούμε. θέρο. Ευχαριστώ. Πολλοί μίλησαν εδώ για την Κίνα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι θύμα κοινωνικού ντάμπινγκ και υπάρχει μεγάλος αθέμητος ε, ανταγωνισμός. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την γεωργία, η οποία πλήττεται στην Ευρώπη, όπως και η χαλιβουργία κατά τη δεκαετία του 70. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει λοιπόν κοινωνική στρέβλωση στον τομέα της γεωργίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την απόσπαση των εργαζομένων και τις ε, κοινωνικές προδιαγραφές, όπου υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός από αυτούς που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δουλέψουν. Jude. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι 80% των εμπορικών συμφωνιών, και δεν είμαι βέβαιη ότι σωστά σημείωσα την ημερομηνία, συμπεριλαμβάνουν και αναφορέ στι βασικέ συμβάσει του ΆΕΛΟ. Υπάρχουν βέλτιστε πρακτικέ από την ε, εφαρμογή όλων αυτών των συμφωνιών και των εργασιακών δικαιωμάτων όπω προβλέπονται από τον ΆΕΛΟ. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τι συζητήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ΣΥΠΑ για την ε, συμφωνία TTIP και για να δούμε τι είδου ε, υλοποίηση των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων θα υπάρξει. Από την οπτική γωνία του αελό, λοιπόν, εσεί πώ το βλέπετε αυτό. Δεύτερη ερώτηση και θα γίνει και ακρόαση για το θέμα του GSP+, το προτιμησιακό καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη του ILO για το θέμα αυτό. Ε, και στο, στη διαδικασία της ανάλυσης συστημικών παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μάλλον με συγχωρείτε, η Επιτροπή για την ε, υλοποίηση των προτύπων χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς για να αποφασιστεί εάν υπάρχει συστηματική παραβίαση των προτύπων του ΑΕΛΟ από κάποιες χώρες ή όχι. Θα έπρεπε να απευθύνουμε έκκληση για λεπτομερέστερη ε, και συστηματικότερη εμπλοκή της Επιτροπής των Επιρογνωμόνων ή να επαφιόμαστε απλώς στην Επιτροπή για την υλοποίηση των προτύπων. Διότι είναι πολύ δύσκολο, όπως ξέρετε, να συμφωνήσουν κυβερνήσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες ανά τον κόσμο για τα θέματα αυτά. Από τη δική σας την οπτική γωνία και γενικότερα επίσης, ξέρουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου βρίσκεται σε δύσκολη θέση πλέον μετά τον Ναϊρόμπι και υπάρχει μια μεγάλη, υπήρχε μια μεγάλη όθηση στο παρελθόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτή τη στιγμή βλέπετε να υπάρχει τάση να ε, μετακινηθούμε προς την διμερή πολυμερή προσέγγιση όπως και στο εμπόριο υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από, από την πολυμερή ή έχετε κάποια άλλη ιδέα. Σας ευχαριστώ. Α, και εγώ λοιπόν να κάνω ορισμένε συμπληρωματικέ ερωτήσει και σχόλια. Ίσως ε, κάπως γενικότερο χαρακτήρα, μιας και πράγματι συζητούμε τη στρατηγική του 21ου αιώνα και εξετάζουμε πού θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και βεβαίως και η κοινή γνώμη εξετάζει εάν όντως η εμπορική πολιτική που ασκούμε βοηθεί ή όχι τον κόσμο, τους ανθρώπους σε αυτό το πλαίσιο παίζουν και τα δικαιώματα των εργαζόμενων πολύ σημαντικό ρόλο. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχουν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Από τη μια μεριά η προώθηση, το, αυτό το promotion των ε, ε, δικαιωμάτων των εργαζόμενων, από την άλλη μεριά η αυστηρή επιβολή τους. Πού νομίζετε, ποιο νομίζετε ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα ή θεωρείτε ίσως ότι πρέπει να ακολουθηθεί μάλλον ένας μέσος δρόμος ανάμεσα σε μια προσπάθεια προώθησης διαφήμισης τους ας πούμε και από την άλλη μεριά επιβολής τους δια όρων που συμπεριλαμβάνουμε, μέσω δηλαδή όρων που συμπεριλαμβάνουμε ε, στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιβολή των προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, μπορείτε να δώσετε κάποια θετικά παραδείγματα γνωρίζουμε το Sustainability Compact, το σύμφωνο βιωσιμότητας του Bangladesh, όπου είπατε και εσείς ότι το μπουκάλι ακόμα είναι μισοάδιο. Είστε ικανοποιημένοι πάντως ε, ως μια αρχή. Ε, θεωρείτε ότι τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, παίξει κάποιο ρόλο. Τρίτο ερώτημα, σε ό,τι αφορά πάλι την εφαρμογή. Η Μαρίτη Σάκ είπε ότι Υπάρχουν χώρες οι οποίες υπογράφουν διάφορες συνθήκες, συμφωνίες του ΑΕΛΟ και δεν τις σέβονται. Ούτως ή άλλως και οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο δύο από τις οχτώ έχουν κυρώσει. Πώς το βλέπετε εσείς, θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμόζονται παρόλο που δεν έχουν περάσει από την φάση της επίσημης κύρωσης. Τέταρτο, και σε άλλες ε, συζητήσεις στρατηγικού χαρακτήρα έχουμε διαπιστώσει ότι σήμερα εξαρτώμεθα πολύ από την παγκόσμια, το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε και όχι τόσο πολύ από την διακρατική διακίνηση εμπορευμάτων. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο σε ό,τι αφορά την προσπάθεια Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Διότι όσο περισσότεροι stakeholder, όσο περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη λοιπόν συνεργάζονται ή συμπλέουν μαζί, τόσο δυσκολότερο γίνεται. Αναφερθήκατε και σε αυτή τη δυνατότητα, αυτό που λέγεται στα αγγλικά name and shame, να κατανομάζονται δηλαδή οι φταίχτες, αυτοί που παραβαίνουν. Μπορώ, αν το αντιστρέψω αυτό, να ρωτήσω αν υπάρχει μια ιδέα για μια πιστοποίηση προϊόντων, εμπορευμάτων, να πιστοποιείται δηλαδή ότι έχουν συμμορφωθεί η παραγωγή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζόμενων κτλ. Τα δικαιώματα των εργαζόμενων στην παραγωγή του συγκεκριμένου είδους. Και το ερώτημα των εμπορικών προτιμήσεων. δεν υπάρχει δυνατότητα και μέσα στο σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων για προϊόντα ή και υπηρεσίες. Όχι δηλαδή συνολικά για μια χώρα, αλλά συγκεκριμένα για ένα είδος παροχής υπηρεσιών. Α, επανήλθε η κυρία Αρενά η οποία ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πολάσκη. Θα ήθελα να κάνω τις ε, εξή παρατηρήσεις. Σε σχέση με το ΔΟΕ και την Δυτική Αφρική, μιλάμε για την φιλελευθερωποίηση της αγοράς, την απελευθέρωση αγοράς που είχε μεγάλες επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά Τώρα μιλάμε για ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Δυτική Αφρική. Θα φροντίσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην εγχώρια αγορά και στις συνθήκες εργασίας. Το δεύτερο θέμα έχει ως εξής. Πόσο προωθήσαμε την αξιοπρεπή εργασία και στις αναπτυγμένες χώρες. Μιλήσατε από 300 εκατομμύρια σε 330 εκατομμύρια και μιλάμε για ε, εργασία στις αναδυόμενες χώρες. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη φτώχεια για τους ε, μισθωτούς. Αυτή όμως η μισθολογική φτώχεια υπάρχει, αφορά και τις αναδυόμενες χώρες, δηλαδή υπάρχει μια φθήνουσα απορία των μισθών στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, διατάξεις σε σχέση με την εργασία οι οποίες να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή σε σχέση με την βιώσιμη εργασία δεν υπάρχουν μηχανισμοί ανταπάντησης για τις χώρες που δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Ως προς την μισθολογική φτώχεια και τα δύο άκρα που υπάρχουν σε αυτό το διάνυσμα θεωρείται ότι υπάρχει μία ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού, ε, πολύ μικρή ποσοστιαία αναλογία η οποία ε, κρατά τον πλούτο στα χέρια της ε, σε αντίθεση με την πολύ μεγάλη και ολοένα διευρυνόμενη φτώχεια. Και μετά από 20 χρόνια ε, συμφωνιών φτάσαμε σε μία κατάσταση όπου η συμφωνία, η συμφωνία ναύτα ε, έφτασε σε, στα επιθυμητά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε σχέση με το Μεξικό. Και ο κύριος Σόλτς καθυστέρησε κάπως όχι κύριε ε, ε, Πρόεδρε δεν καθυστέρησα, απλώς δεν σημειώσα το όνομά μου προηγουμένως. Σας ευχαριστώ κυρία Πολάσκη. Τρεις ερωτήσεις που νομίζω δεν έχουν τεθεί. Στην κοινή δήλωσή σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνεται ότι και το μεταναστευτικό αποτελεί σημαντική πρόκληση. Και μιλούμε άλλωστε και για τη διασύνδεση εδώ και με το διεθνές εμπόριο και με τον ρόλο του ε, Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Εμπορίου. Αναφέρεστε και στη συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δούμε όμως την πραγματικότητα από τις αρχές του έτους, μάλιστα από τον προηγούμενο Οκτώβριο, η κατάσταση έχει γίνει δραματική. Με ενδιαφέρει τώρα να μάθω αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή και ILO που εντοπίζεται στις δυνατότητες προοπτικής απασχόλησης και στην ισότητα αμοιβών ανάμεσα σε απασχολούμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε αυτούς που έρχονται απ' έξω. Δεύτερο που με ενδιαφέρει υπάρχει και μια αύξηση της ανισότητας στα εισοδήματα αλλά και στους μισθούς και στις αμοιβέ. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις γυναίκες. Πώς μπορεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΑΕΛΟ να επηρεάσει την πορεία αυτή προς κάτι προς μια καλύτερη κατεύθυνση για να μειωθούν οι ανισότητες. Θα αρκεστώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Με ενδιαφέρει όμως το ερώτημα εάν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε δεσμευτική την εφαρμογή των προτύπων του ΑΕΛΟ όταν μιλούμε για διεθνείς συμφωνίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν κεφάλαιο βιωσιμότητας που να περιλαμβάνει και κριτήρια απασχολησιμότητας και που να είναι δεσμευτικά ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών των τρίτων χωρών. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πολάσκη, σας επιστρέφω το μικρόφωνο. Έχετε πολλές ερωτήσεις που καλείστε να απαντήσετε. Και μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα μπορέσει να αντιδράσει στα όσα θα πείτε εσείς. <laughs> I didn't know, but now I know I have time enough. So um, a number of the questions Ευχαριστώ πολύ. Πλήθο ερωτήσει, αλλά θα προσπαθήσω. Κάποιε άλλωστε καλύπτουν το ίδιο θέμα λίγο πολύ. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να πάω και χρονικά πίσω στις παρεμβάσει. Οι πιο πρόσφατε είναι αυτές που μείναν και πιο πολύ στο νου. Το θέμα της μετανάστευση, λοιπόν πρώτα απ' όλα. Ο ΑΕΛΟ ασχολείται πολύ με τα θέματα μετανάστευση, ιδίω για την νόμιμη μετανάστευση. Συζητούμε ήδη με πολλέ χώρε για να δούμε τι διμερείς ή πολυμερείς διαπραγματεύσεις μπορεί να έχουν με μεταναστευτικές συμφωνίες και εφόσον υπάρχουν και εμπορικές διατάξεις αυτές. Έχουμε κοιτάξει λοιπόν ήδη τι υπάρχει και πριν την τεράστια ε, έξοδο μεταναστών από τη Συρία στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Όμως ήδη υπήρχαν ε, τάσεις μετανάστευσης και στη Μέση Ανατολή και στην Νότια Ανατολική Ασία. Οπότε κοιτάζουμε οι συμφωνίες μετανάστευσης να προβλέπουν τουλάχιστον ένα δίκτυο βασικής προστασίας στη φάση της πρόσληψης, της ε, διέλευσης και του τι είδου υποδοχή θα λάβουν από τις χώρες υποδοχής. Και αυτό για να υπάρχουν συνθήκες ε, αξιοπρεπούς εργασίας, η αποφυγή της εκμετάλλευσης ή δυνατόν και της διακίνησης ή εμπορίας ανθρώπων. Θέλουμε βασικά να υπάρχει προστασία και κάποια βεβαιότητα για τα εργασιακά πρότυπα στη χώρα υποδοχής. Εάν οι μετανάστες είναι απελπισμένοι φτάνοντας σε μια χώρα, θα, ε, και δεν υπάρχουν τα επαρκή εργασιακά πρότυπα, θα εργαστούν όπως να είναι ε, και σε συνθήκες επισφάλειας και ανασφάλειας προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Υπάρχει λοιπόν εντατική συνεργασία με πολλές χώρες και τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρωθεί ακριβώς στις βασικές συμφωνίες που ήδη ισχύουν. Έχουμε συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό νομίζω ότι επιτείνεται τώρα ως μορφή συνεργασία λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση δεν θέλω να πω με αύξηση, θα έλεγα περισσότερο με έκρηξη της μετανάστευσης, Οπότε ασχολούμαστε πολύ με το διάλογο Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική, Αφρικανική Ένωση για τη μετανάστευση, μετανάστευση μεταξύ των δύο υπήρων και ε, να δούμε κατά πόσο μπορούν να βελτιωθούν οι όροι της μετανάστευσης αυτής. Επίσης, στο βαθμό που είναι δυνατό αυτό, ασχολούμαστε και με την ε, ε, προσπάθεια να δημιουργηθούν θέσει εργασία στι χώρε που είναι εκείνε οι οποίε στέλνουν μετανάστε αλλού. Λόγω τη πολιτική του αστάθεια, λόγω κάποιων εχθροπραξιών που μπορεί να μην έχουν επιληθεί. Είμαστε λοιπόν πολύ δραστήριοι στη συνεργασία μα με την Τουρκία, την Ιορδανία και άλλε χώρε, προσπαθώντα να δημιουργήσουμε προγράμματα απασχόληση που μπορεί και να απορροφήσουν του μετανάστε, του ενδυνάμει μετανάστε, αλλά να δημιουργήσουν και δυνατότητε για του ε, μη απασχολούμενους, ε, εγχώριους εργαζόμενους. Όπως έχει δείξει πείρα μας από την Ευρώπη, αν υπάρξει μια εισρωή 2 εκατομμυρίων από την Τουρκία λόγου χάρη, εκ των οποίων 800.000 θέλουν να εργαστούν ε, και μπορεί να είναι και περισσότεροι, εάν δημιουργηθούν θέσει απασχόληση για εκείνου, αλλά είναι πολύ άνεργοι ή μη απασχολούμενοι στην Τουρκία, σε τουρκικέ οικογένειε, τα πράγματα θα είναι άσχημα. Έχουμε κάποιες, ε, κάποια παραδείγματα από καλά προγράμματα μικρή κλίμακα, αλλά για να γίνει αυτό σε μεγαλύτερη εμβέλεια χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ε, χρήση πόρων. Ε, μπορεί να υπάρξουν αμέσω όμω αυτοί οι πόροι. Υπάρχει ανάγκη υποδομών, υπάρχει ανάγκη για δρόμου και λιμάνια, νοσοκομεία. Ε, για δημοτικά σχολεία. Σε πολλέ λοιπόν περιπτώσει με χρηματοδότηση αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, αλλά απαιτούν πολύ εντατική εργασία, είναι πολύ εντατικά από την άποψη του δυναμικού που αποσχολούν. Πρόσφατα, μια εβδομάδα νομίζω την Κυριακή, συμμετείχα σε μια διάσκεψη στο Λονδίνο που εξέφρασα κάποιε πολύ συγκεκριμένε ε, προτάσει. Ήταν εκεί κι άλλοι ηθήνοντε και ελπίζω η στήριξη να υπάρξει. Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει λοιπόν ο ΑΕΛΟ. προσπαθούμε, ε, συμμετέχουμε ενεργά, αλλά πρέπει να υπάρχει καλό συνδυασμό με του πολιτικού ευθύνοντε για το σωστό σχεδιασμό πολιτικών. Για να δημιουργηθούν στην πράξη εργασιακέ ευκαιρίε και να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Η ερώτηση για την Δυτική Αφρική. Πρέπει να πω ότι ο οργανισμός μας παράγει μια σωρία εκθέσεων. Δεν ξέρω σε ποια αναφέρεστε πολλούς αλλά για τα εμπορικά ανοίγματα τη Δυτική Αφρική και κατά πόσο αυτά είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ανεργία. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να απαντήσω γενικότερα ε, και όχι συγκεκριμένα για αυτή την περιοχή του κόσμου. Όσοι μελετούν την εργασία σε αυτέ τι περιπτώσει χρησιμοποιούν κάποια μοντέλα, τα λεγόμενα μοντέλα τη Ευρωπαϊκή όπω ονομάζονται, και βλέπουν στη δομή τη οικονομία πώ οι εμπορικοί εταίροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιε εκτιμήσει γιατί ε, μπορεί να αλλάξουν οι οικονομικές εξελίξεις εφόσον ε, περιοριστούν κάποιοι εμπορικοί φραγμοί λόγου χάρη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις όπου κάποιες χώρες έχουν περίπου το ίδιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ξεκινούν ε, μια συμφωνία, μια συνεργασία εμπορικής απελευθέρωσης όπου εκεί ο αντίκτυπος είναι θετικός. Δυστυχώ τα μοντέλα όμω αυτά μέχρι πρόσφατα ε, βασίζονται στην εικασία ότι υπάρχει πλήρη απασχόληση και ότι όλοι θα άλλαζαν θέση εργασία, αλλά κανεί δεν θα έμενε χωρί ε, καρέκλα όταν θα σταματούσε αυτό το παιχνίδι. Ε, έτσι μπορεί να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, όταν οι χώρε είναι και δύο προηγμένε, χώρε υψηλού εισοδήματο, υπάρχουν σοβαρέ πιθανότητε, υπάρχει μια ουδέτερη ανασύνθεση τη εικόνα τη απασχόληση δηλαδή μια πολύ βραδία εξέλιξη του βιωτικού επίπεδου με πολύ μικρό θετικό αντίκτυπο, αλλά κάποιε φορέ υπάρχουν και δυσμενεί επιπτώσει. Αυτό συνέβη στην, στο Μεξικό μετά τη Συμφωνία Ναύτα. Εκεί μια οικονομία που είχε ένα πολύ μεγάλο γεωργικό κλάδο με πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Δηλαδή πολύ περισσότεροι απασχολούνταν από ότι η αξία που παρήγαν και που προσέφερε ο κλάδος αυτό στην οικονομία της χώρας. Άνοιξαν σε μια οικονομία που ήταν πιο αποτελεσματική στον κλάδο της γεωργίας, πριν δημιουργήσουν θέσει απασχόληση στι υπηρεσίε και την κατασκευή. Οπότε για πολύ μεγάλο διάστημα υπήρξε αρνητικό αντίκτυπο για την απασχόληση. Είδαμε λοιπόν τι ε, επιπτώσει είχε αυτό για το Μεξικό. Παρόλο που κάποια στιγμή οι οικονομίε προσαρμόζονται, δεν μένουν έτσι σταθερά και σε τέλμα τα πράγματα για πάντα, όμω είναι πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά. Και όπω είπα, στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε τι προβλέψει μα και τα μοντέλα στα οποία βασιζόμαστε, βασιζόμαστε στην ενοικασία ότι υπάρχει πλήρη απασχόληση και στι δύο χώρε. Ε, εάν μελετήσει κανεί πιο συγκεκριμένα την απασχόληση όμω, μπορεί να δει ότι, ε, ότι με και μεσοπρόθεσμα από τι συμφωνίε αυτέ προκύπτουν και αρνητικέ επιπτώσει. Για να επανέλθω στι ερωτήσει του κυρίου Λάγκε. Το ερώτημα για τη φιλοσοφική μα προσέγγιση και το κατά πόσον θέλουμε να υπάρχει προώθηση των βελτιωμένων εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών ε, συνθήκων και το κατά πόσον προβλέπονται σχετικέ κυρώσει. Ε, εάν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος για να καταγράφουμε και να ανταμείβουμε τις καλές επιδόσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση η πρόθεση αυτών των προτύπων να μην είναι θετική. Πάντοτε υπάρχει κάτι να μάθει κανεί, υπάρχουν καλέ πολιτικέ που πρέπει κανεί να μελετήσει, να προσαρμόσει, να μιμηθούν άλλε χώρε. Η προώθηση λοιπόν είναι πάντοτε η βέλτιστη λύση. Όμω αυτό που θα έλεγα για τι κυρώσει είναι ότι κατά πρώτον δεν θα χρησιμοποιήσω αναγκαίο τον όρο ε, κυρώσει, αλλά αποτροπή περισσότερο. Διότι όταν οι εμπορικέ συμφωνίε λόγω χάρη δημιουργούν το δυναμικό να μην αντληθούν ωφέλη εφόσον οι εταίροι δεν υλοποιούν πλήρω τι υποχρεώσει που είχαν αναλάβει ε, συνάπτοντα τη συμφωνία τα μέρη δηλαδή συμφώνησαν να κάνουν κάτι και το αποτέλεσμα θα είναι και οι δύο να λάβουν ωφέλη, αλλά όταν κάποιο δεν φέρει πέρα όλε τι υποχρεώσει, ο άλλο αφήνει τα εργασιακά κατά μέρο προ στιγμή και βάσει των υπόλοιπων εμπορικών ρητρών μπορεί να αποσυρθεί από τα υπόλοιπα ωφέλη που θα αποκόμιζε ε, ανάλογα με τη συμπεριφορά του εταίρου. Αυτού του είδους η αποτροπή πρέπει να ε, εφαρμοστεί και για την βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και ε, στην στο σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν μπορεί να βασίζεται στην ερμηνεία των ρητρών για τα εργασιακά δικαιώματα. Αν κάποιο δεν φέρνει πέρα όλε υποχρεώσει του, ο άλλο μπορεί να αποσυρθεί. Και θα μπορούσε κανεί τι εργασιακέ ρήτρε να τι έχει σε πολύ ε, χαμηλότερο επίπεδο από ότι τις οικονομικές ρήτρες μιας συμφωνίας. Τα πάντα εξαρτώνται από αυτό. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να υπάρχουν κυρώσει στι εμπορικέ ή οποιασδήποτε άλλε συμφωνίε. Η αποτροπή πιστεύω ότι είναι ο καλύτερο τρόπο θετικά να δοθούν κίνητρα για την συμμόρφωση, αλλά ταυτόχρονα η προώθηση, όπω είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρο τη όλη προσπάθεια. Εάν υπάρχουν θετικές προσεγγίσεις έω τώρα. Νομίζω σα έδωσα ένα-δυο παραδείγματα από καλά εργασιακά προγράμματα σε χώρες που αφορούν 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενου, όπου η παρακολούθηση από τη δουλειά στα εργοστάσια και τα αποτελέσματα της συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Πρώτα απ' όλα γίνεται απόρριτα μεταξύ εργοστασίου και υπευθύνου και μετά δημοσιοποιούνται μόνο αν δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματα ακόμη και αν έχουν επιληθεί, τότε δημοσιεύονται ω θετικό παράδειγμα. Αυτό, κύριε Λάγκε, νομίζω ότι απαντά στην ερώτησή σα για την επισήμανση. Εάν οι πληροφορίε που προκύπτουν είναι αρκετά ακριβεί, τότε δεν υπάρχει λόγο να λάβει κανεί δράση. Ε, δηλαδή, ε, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο τομέα. Ξέρουμε για ποιον τομέα μιλάμε, αλλά δεν μπορούμε να το ε, κάνουμε συγκεκριμένο σε επίπεδο εργοστασίου. Εκεί πρέπει να είναι κανεί πολύ ακριβή, να προσέχει για το αν μιλάει για ένα εργοστάσιο 500 ή 20.000 εργαζομένων. Εάν υπάρχει το όνομα του εργοστασίου και μπορεί να το, κατανο... να το καταδείξει κανείς στην πράξη. Οι πληροφορίες λοιπόν πρέπει να είναι αξιόπιστες, πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί από ε, εκπροσώπους ή υπευθύνους που δεν έχουν καμία σύγκρουση συμφέροντος, πρέπει να, είναι, να έχουν κύρος, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει τον έλεγχο να ξέρουν ποια είναι ακριβώς τα πρότυπα και τι είδους συμμόρφωση απαιτείται. Γι' αυτό έχει πετύχει αποτέλεσμα το ΕΛΟ με το σύστημα καλύτερη εργασία, γιατί ακριβώς όλοι γνωρίζουν τα πρότυπα του ΕΛΟ και φροντίσαμε να, να προσλάβουμε υπευθύνου που δεν είναι διεθνεί εργαζόμενοι με διεθνεί υψηλού μισθού, αλλά εργάζονται τοπικώ και κοιτάζουν την τοπική πραγματικότητα πιο κοντά. Αυτό μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα, θα μπορούσε να επαναληφθεί σε πολλού άλλου κλάδου. Έχουμε πολλέ αναπτυσσόμενε χώρε που έρχονται στον ILO και λένε παρακαλούμε το πρόγραμμα Better Work, εφαρμόστε το στα μα εργοστάσια και μπορεί αυτέ οι χώρε να συμμετέχουν όντω στι διεθνεί αλυσίδε προμήθεια, στι global supply chains όπω έχουμε ονομαστεί. Αυτά λοιπόν όλα είναι σημαντικά γιατί και οι αγοραστέ και αυτοί που πολλούν και αγοράζουν βρίσκουν ότι έχουν αξία και προστιθέμενη αξία αυτά τα προγράμματα τα συστήματα αυτά από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να ε, μπορούν να σταθούν μόνα του. Αλλά στην αρχή χρειάζεται μια παρέμβαση από δική μα πλευρά. Υπάρχουν και πολλέ άλλε ερωτήσει για το κατά πόσον η κύρωση των συμβάσεων ε, συνάδει με την εφαρμογή των συμβάσεων. Δηλαδή, εάν στην πράξη υπάρχει ανάλογη ανάληψη υποχρεώσεων. Για τις βασικές μας συμβάσεις, τι να σας πω, εγώ είμαι ε, αξιωματούχος του ILO, δεν μπορώ να σας, πω παρα, ε, να σας απαντήσω παρά καταφατικά. Οι χώρες καλώς κυρώνουν τις συμβάσεις του ILO, δηλαδή μιλάμε για βασικά δικαιώματα, προστασία των παιδιών από την εργασία, από την καταναγκαστική εργασία, μη διακριτική μεταχείριση, ελευθερία του συνασπίζεστε και του, ε, και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά με την δήλωση του 1988 που θεσπίζει αυτά τα βασικά εργασιακά πρότυπα, ε, και που θα ισχύουν για όλες τις χώρες ασχέτως κύρωσης ή όχι, είναι πραγματικά ένα ορόσημο, είναι μια καμπή στην όλη προσέγγιση του έλου. Διότι ε, είτε μια χώρα έχει κυρώσει είτε όχι τη σύμβαση, καλό να το κάνει βέβαια, αλλά είτε συμμετέχετε είτε όχι στον ΕΛΟ, αφού ανήκει στη διεθνή κοινότητα, αναλαμβάνει κάποιες υποχρεώσεις, μια και έχει οικονομικές δραστηριότητε σε αυτή τη διεθνή κοινότητα. Έχει την υποχρέωση να σέβεται αυτές τις βασικές υποχρεώσεις. Αυτό το συμφώνησαν τα 148 κρατη μέλη μας με κάποιες μικρές εποχέ, με κάποιε χώρε που ξέραν ότι τα εργασιακά του δεν είναι τόσο καλά, αλλά συντριπτικά η πλειοψηφία, το 95% των χωρών, καθώ και οι ενώσει των εργοδοτών και των εργαζομένων, υπερψήφισαν αυτή την προσέγγιση. Είναι λοιπόν ένα διεθνέ πρότυπο. Αυτά τα τέσσερα εργασιακά βασικά δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται σε όλε τι συμβάσει και ότι εφαρμόζονται σε όλε τι χώρε ασχέτω τη ε, κύρωση ή όχι. Οπότε ναι, από τη μια όλε οι χώρε θα κυρώσουν τι συμβάσει, θα το έλεγα, αλλά από την άλλη υποχρεώσει έτσι κι αλλιώ υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται. Από την πλευρά του συστήματο εποπτεία του ILO, ε, οι χώρες που έχουν κυρώσει τις συμβάσεις περνούν μια διαδικασία συστηματικότερη και θα έλεγα και λίγο πιο αυστηρή από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για το κατά πόσον συμμορφούνται ή όχι. Οι χώρες αξιολογούνται όλες για τα εργασιακά ε, πρότυπα, ασχέτως κύρωσης. Όμως ε, υπάρχει ένα κύκλος τετραετίας, δηλαδή δεν γίνεται αναετήσιο βάση η εποπτεία αυτή στις χώρες που δεν έχουν κυρώσει, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρή. Αυτό δεν τι απαλλάσσει πάντω από τι ευθύνε του βάσει των εμπορικών συμφωνιών, γιατί είναι υποχρεωμένε να σέβονται τα βασικά εργασιακά πρότυπα. Η, η επικοινωνία είναι προφανώ ένα ε, πολύ βασικό θέμα η εφαρμογή είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν αρκεί ένα σύστημα όπου υπάρχουν μόνο θεωρητικές υποχρεώσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει υλοποίηση από τις κυβερνήσεις, πρακτική εφαρμογή, διότι κανείς και ο θελός δεν μπορεί να συμμορφούται και πρέπει να υπάρχει και αποτροπή, όπως έλεγα προηγουμένως, όχι αναγκαστικά κυρώσεις, για να βεβαιωνόμαστε ότι ο σεβασμός προκύπτει. Και μετά υπάρχουν και τα εργασιακά πρότυπα. Δεν χρειάζεται να σας πω, μπορείτε να ανοίξετε τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και μέσα σε μια εβδομάδα θα δείτε εικόνες και βίντεο από χώρε που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα παντού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και απαντά και σε κάποιε από τι υπόλοιπε ερωτήσει που τέθηκαν. Δηλαδή, εάν αυτή η ενοποίηση τη παγκόσμια ε, οικονομία θα βελτίωνε τα εργασιακά πρότυπα. Σε κάποιε περιπτώσει συνέβη αυτό. Υπήρξε πίεση προ τα πάνω σε πολλέ χώρε να βελτιώσουν τα εργασιακά του πρότυπα. Όμω, όχι μόνο οι εμπορικέ συμφωνίε, ούτε καν απλώ οι γενικέ πιέσει τη παγκοσμιοποίηση, αλλά και άλλε δυνάμει έχουν συμβάλει στην εξέλιξη τη φτώχεια. Ξέρουμε όλου του αριθμού. Εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπων έχουν ξεφύγει από τη φτώχεια από τότε που εγκρίθηκαν οι στόχοι τη χιλιετία ε, του ΟΗΕ. Ε, οι περισσότεροι ήταν στην Κίνα. Εάν δεν συμπεριλάβουμε την Κίνα σε αυτόν τον υπολογισμό, δεν θα είχαμε πετύχει το στόχο ε, σχετική καταπολέμηση τη φτώχεια μέχρι το 2015. Τα πράγματα θα είχαν ε, πάει πολύ χειρότερα. Δεν θα υπήρχε λοιπόν αυτή η βασική βελτίωση, αλλά τελικά υπήρξε. Και αυτό απαντά και σε κάποιε από τι υπόλοιπε ερωτήσει που τέθηκαν ούτω ή άλλω και τις οποίες θα επανέλθω. Νομίζω το κατονομάζει και επωνυθίζουν το κάλυψα. Τώρα το θέμα της επισήμανσης, του κατά πόσον μπορούμε να βάλουμε ένα σήμα πάνω σε αυτούς που ε, έχουν κάνει κάποια παραβίαση ή όχι. Είναι και θέμα το πόσο ακριβής είναι, ε, το πόσο ακριβής είναι Ε, για την Κίνα τώρα. Ε, ο ILO δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση γι' αυτό. Πολλοί, όπω η Κίνα και άλλοι που εκπροσωπούν χώρε που είναι μέλη του ILO εδώ σε αυτή την αίθουσα, ε, έχουν αυτέ τι υποχρεώσει, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε θέση, ε, διότι δεν εκπροσωπούμε αυτή τη σκοπιά του θέματο. Τώρα για το τι γίνεται για τα εργασιακά ε, και το Ιράν. Υπήρξαν παράπονα από καιρού καιρών για θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, όχι το Ιράν. Και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές και ε, χρηματικές κυρώσεις έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε χρηματικές συναλλαγές ε, ούτε μπορούμε να έχουμε τέτοια παρουσία ή πίεση προς το Ιράν όπως κάναμε κάποια, κάποτε στο παρελθόν. Ίσως να ξαναπροκύψει στο μέλλον αυτή η δυνατότητα. Νομίζω μιλήσαμε αρκετές φορές για την κύρωση. Κάποιος με ρώτησε εάν τα προγράμματα της Ένωσης είναι, το πρόγραμμα της Ένωσης είναι παρκώς φιλόδοξο. Νομίζω ότι πλήρωνες βουλευτέ με ρώτησαν το πράγμα αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά που πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά κοινωνικά, ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και στο διεθνές σύστημα και συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνει σε συγκεκριμένες συμφωνίες είτε εξετάζεται συγκεκριμένα μέτρα ad hoc όπως το σύμφωνο με τον Μπάγκλαντες Νομίζω ότι η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων εκείνων προσπαθούν να επιφέρουν κάποια πρόοδο και αυτό είναι καλά νέα, πολύ καλά νέα, αυτά αποτελούν πολύ καλά νέα δηλαδή. Και συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες, αλλά η επιτυχία των προσπαθειών απέναντι στο μέγεθος των προκλήσεων σαφώς υπολείπονται οι προσπάθειες οι νέε στρατηγικέ και η δουλειά που κάνει η δική σα Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αποτελούν και μια σιωπηρή αναγνώριση ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα. Πάντω έχουν επιτευχθεί ορισμένα πράγματα και δείχνουν να πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίω χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τα προβλήματα που σημειώνονται στι παγκόσμιες αλυσίδε παραγωγή σε ε, χώρες εταίρους, ιδίως ε, του τρίτου κόσμου, Χρειάζεται βεβαίω να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Μίλησα και για το ζήτημα της προώθησης των προτύπων του ILO ή της εφαρμογής του μέσω, της εφαρμογής τους, της επιβολής τους μάλλον, μέσω όρων στις ε, συμφωνίες. Αν προσπαθήσω να απλοποιήσω κάπως την εικόνα, θα μπορούσα να πω ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον πιο φιλόδοξες από αυτές που επιβάλλουν οι Ενωμένες Πολιτείες. Η δημιουργία αποτροπής μέσω του ελέγχου είναι μάλλον πιο ισχυρή από την πλευρά των Αμερικανών. Μπορεί ίσως να καταλήξει κανείς σε μια ε, συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις που να είναι η καλύτερη δυνατή και να είναι αμοιβαία αποφελής. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχετε μπροστά σα σε ό,τι αφορά την εποπτεία των διαπραγματεύσεων αυτών. Μια μηδέα εποφελής έκβαση θα πρέπει να μετρηθεί σε επίπεδο παγκόσμιο. Και άλλε χώρε τότε θα οδηγηθούν να προσπαθήσουν να συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτού του επίπεδου. Βεβαίω υπάρχει μεγάλη συζήτηση ακόμη για το, πού βρισκόμαστε και πού μπορούμε να καταλήξουμε. Τώρα το ερώτημά σα για, το κοινωνικό dumping και ιδίω ό,τι αφορά την γεωργία και τι ε, κοινωνικέ συνθήκε απασχόληση των εργαζόμενων στην γεωργία. Αυτό παραπέμπει στο θέμα που ανέπτυξα σχετικά με τη συμφωνία ναύτα με το Μεξικό. Όταν έχετε, όταν υπάρχει ένα άνοιγμα στι οικονομικέ σχέσει μέσω μια εμπορική συμφωνία. και υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα και εισοδήματος και παραγωγικότητας και ικανοτήτων και επίπεδου ζωής μεταξύ των δύο μέρων, των δύο χωρών. Θα υπάρξουν βεβαίως, θα απορρεύσουν από αυτά κάποιες συνέπειες που δεν είχατε την πρόθεση να επιτύχετε. Θα υπάρξει κάποια σύγκληση βέβαια σε μια τάση να ανυψωθεί το επίπεδο, θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η σύγκριση θα γίνει οπωσδήποτε προς τα πάνω. Χρειάζεται λοιπόν να λαμβάνετε πάντα υπόψη αυτό. Αυτό μπορεί να απαιτήσει και κάποια υποστήριξη στην ανάπτυξη με μεγαλύτερη συνεργασία για παράδειγμα και εκτός εμπορικών συμφωνιών. Πάντως δεν θα ήθελε κανείς οι εμπορικέ συμφωνίες που συνάπτει να οδηγήσουν σε μια σύγκληση προς τα κάτω. Είναι όμως υπαρκτό ο κίνδυνος αυτός. Όταν είπα στην αρχή της ομιλία μου ότι οι σύγχρονε πτυχές της παγκοσμιοποίηση έχουν σχέση με αυτή την τεράστια προσφορά εργατικού δυναμικού μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου με την Κίνα που μπαίνει στο παιχνίδι της παραγωγής δεν υπήρξε σύγκριση προς τα κάτω, υπήρξε σύγκριση προς το μέσον. Δηλαδή έχει σηκωθεί το κάτω γιατί η Κίνα αύξησε τους κατώτατους μισθούς σε τεράστιο ποσοστό την τελευταία δεκαετία. Επομένως σύγκριση προς τα πάνω. Και όμως είδαμε και μείωση των απολαβών σε αναπτυγμένες οικονομίες. Βεβαίως και το είδαμε και αυτό. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό οφείλεται στην παγκόσμια οικονομική ενοποίηση. Ναι, υπάρχει, υπάρχει και αυτό. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και η τεχνολογική ανάπτυξη και εξέλιξη. Έτσι λοιπόν επανέρχομαι στο θέμα των διαπραγματεύσεων και τον σχεδιασμό της πολιτικής. Αν επιθυμείτε να αποφύγετε αυτόν τον ανταγωνισμό προς μια μέση, ένα μέσο επίπεδο, πρέπει να λάβετε μέτρα και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες ανεπτυγμένου εισοδήματος. Μου έγινε και μια εξειδικευμένη ε, ερώτηση για τις γενικευμένες προτιμήσεις και αν αυτές θα πρέπει να βασίζονται μοναχά στην εφαρμογή των προτύπων. Κατά τη γνώμη μου, η αδίποτε τέτοια πολιτική, GSP GSP-SYN για παράδειγμα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλο το εποπτικό έργο του ILO. Έχουμε την γνωστή αυτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ε, περιλαμβάνει εμπειρογνωμοσύνη από πολλές χώρες, πολλές γλώσσες και ούτω καθεξής και μάνατζερ οι οποίοι συνέρχονται για να συζητήσουν πώς θα εφαρμοστούν οι συνθήκες αυτές στις συγκεκριμένε καταστάσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση ή προς την εσφαλμένη κατάσταση. Ε, τεράστιος πλούτος. Πρέπει να γνωρίζετε βέβαια και τη γλώσσα στην οποία σημειώνει η εν λόγω Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ότι κάτι δεν πάει καλά ή πρέπει να δείτε δηλαδή και τις διατυπώσεις που χρησιμοποιεί όταν λέει για παράδειγμα χαιρετίζει με ενθουσιασμό σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά χαιρετίζει απλά σημαίνει ότι τα πράγματα είναι μέτρια και ούτω καθεξής χρειάζεται λοιπόν να εποφεληθείτε και από τον πλούτο των γνώσεων που διαθέτει ο ΑΕΛΟ τέλος ο ΑΕΛΟ μετέφερε την προσοχή του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις πολυμερείς συμφωνίες προς τις διμερείς. Όχι, εμείς εδώ ακολουθούμε. We follow the crowd. Δεν παίζουμε ηγετικό ρόλο. Εφόσον αλλάζει η τάση, ακολουθούμε και εμείς. Όπως φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσά πιστεύουμε ότι πολυμερεί συστήματα προσφέρουν πλονεκτήματα σε όλες τις χώρες και έχουν λιγότερες σε επιπτώσεις από διμερείς Κύριε Πρόεδρε, αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην κυρία Τούνιγκα, που είναι επικεφαλής του τμήματος εμπορίου και βιωσιμότητας στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Είστε μάλιστα η νέα διευθυντή, δεν είναι. Και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μας καλέσατε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σας ευχαριστώ γιατί καταβάλατε κάθε προσπάθεια να προφέρετε καλά το, ή σωστά μάλλον, το όνομά μου. Ε, βρίσκομαι στη θέση αυτή από την 1η Ιανουαρίου. Δυστυχώς πρέπει να ταξιδέψω σε μια μισή ώρα, γι' αυτό αύριο δεν θα παρευρίσκομαι στη συζήτηση για θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητάς μου και που θα συζητηθούν αύριο. Σε σχέση με τα λεγόμενα της κυρίας Πολάσκη θα ήθελα να πω ότι κάνουμε πολλά από κοινού είμαστε σε εβδομαδιαία βάση σε επαφή με το ILO. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή συνεργασία που μας βοηθά και στο δικό μας έργο. Πολλά θέματα που συζητούνται εδώ σχετίζονται με τις εμπορικές συμφωνίες. Αύριο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι οι διατάξεις για την εργασία είναι δεσμευτικές και έχουμε έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Είπατε κυρία Πολάσκη ότι οι συμφωνίες των ΗΠΑ δεν είναι τόσο φιλόδοξες σε σχέση με τις ε, δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές ε, διατάξεις, ιδιαίτερα για την επίλυση διαφορών. Μιλήσατε για τις ε, προτιμήσεις, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων Plus θα συζητηθεί αύριο για τη νέα μας εμπορική στρατηγική τώρα. Πιστεύω ότι θα μας δώσει νέες δυνατότητες για να ασχοληθούμε με την αξιοπρεπή εργασία και άλλα συναφή ζητήματα σε σχέση με την ε, ε, αλυσίδα προμηθειών. Όπως ξέρετε, ε, αύριο θα συζητήσω αυτό το θέμα, γιατί δεν προσδίδει μόνο η Κομισιόν Σημασία στο θέμα, αλλά και τα κράτη-μέλη. Έχει μεγάλη σημασία στην εμπορική μας στρατηγική και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ακριβώς διότι οι παγκόσμιες αυτές αλυσίδες θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα του ILO και στη νέα διάσκεψη, ιδιαίτερα για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Χρησιμοποιούμε αυτά τα εμπορικά μέσα για να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με τις, ε, ε, με τις χώρες εταίρους όχι μόνο στις εμπορικές συμφωνίες, μιλήσατε για τον Bangladesh Compact, αυτό το σύμφωνο με το Bangladesh, όπου συμμετέχει και ο ιδιωτικός ε, τομέας. Νομίζω το ILO γνωρίζει πολύ καλά πόση προσπάθεια έχει καταβληθεί. Μια τρίτη χώρα θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε αυτό το πλαίσιο γιατί είναι μια επίπονη εργασία με τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Και συνεργαζόμαστε και με τις ΗΠΑ και τον Καναδά για το σύμφωνο του Μπαγκλαντές. Χρειάζεται να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες, ίσως το ποτήρι να μην είναι πάντα γεμάτο, αλλά πρέπει να καταβάλουμε τις προσπάθειές μας. Όπως γνωρίζετε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια ε, της διεθνούς συνεργασίας με το ΔΟΕ, τον ΟΣΑ, που ασχολείται ακριβώς με αυτές τις ε, αλυσίδες προμηθειών και ως προς τις βασικές συμφωνίες έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία να τηρηθούν και έχουμε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας με το ΔΟΕ. Έχουμε πολλές ε, πρωτοβουλίες λοιπόν. Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ε, ένα συγκεκριμένο έργο. Συνεργαζόμαστε όχι μόνο με το ILO και τον ΝΟΣΑ, αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα σας αποβάλω μία ερώτηση, κυρία Τουνίγκα. Έχουμε πολλές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στο τομέα της ε, κλωστοϊφαντουργίας. Μιλήσατε για το σύμφωνο με το Μπαγκλατέσκια. και υπάρχει μια φήμη ότι υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν. Την ακούμε εδώ και καιρό. Ότι υπάρχουν ε, ομάδες εργασίας δηλαδή. Αυτή η πρωτοβουλία γκάμιτ θα προωθηθεί και μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με το ILO. Πολλά μου ζητάτε. Η Γενική Διεύθυνση που ασχολήθηκε με αυτό το τομέα είναι μία άλλη Γενική Διεύθυνση. Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει το θέμα της ε, κλωστοϊφαντουργίας και ένδυσης που απασχολεί την ε, Γενική Διεύθυνση Τεύκο και ε, υπάρχει ένα σχέδιο να ασχοληθούμε και με τον τομέα της ένδυσης και της κλωστοϊφαντουργίας. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα συγκλίνουν τα πράγματα ε, Συνεργαζόμαστε με το ΔΟΕ, τον ΟΣΑ, για να δούμε τι ε, ε, συνεργασία υπάρχει σε αυτό το τομέα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας δώσουμε μία συναφή απάντηση ως Κομισιόν. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προς την κυρία Πολάσκη τώρα μία ερώτηση. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση των δικαιωμάτων εργασίας. Πολλές χώρες προσπαθούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται, οι ιδιωτικές εταιρείες. Πώς μπορείτε να συντονίσετε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες, πώς μπορείτε να προβείτε στο συντονισμό. ILO. Ναι, αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή το θέμα του συντονισμού Γνωρίζετε ότι μεταξύ κρατών μελών και βιομηχανικών τομέων υπάρχει πρόβλημα ε, συντονισμού που είναι πολύ χρονοβόρο. Υπάρχει ε, ανταγωνισμός ε, από τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά εν πάση περιπτώσει οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι πολύ μεγάλες για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και επειδή έχω ασχοληθεί 40 χρόνια με το θέμα, ε, δεν μπορώ παρά να καλωσορίσω τις πρωτοβουλίες, διότι δεν θα είναι όλες επιτυχείς, αλλά χρειάζονται όλο ένα και περισσότερες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, όπως είπε και η κυρία Τουνίγκα. Δηλαδή χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες για να κάνουμε τη διαφορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές τις πρωτοβουλίες για να υπάρχει καλός συντονισμός. Θα πρέπει να υπάρχει και μετριοφροσύνη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε μία αξιολόγηση για να δούμε πού υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και πού είναι πραγματικά παραγωγικά. Γιατί δεν έχουμε πάντα τους πόρους και τις ικανότητες. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού. Επίσης, όπως γνωρίζετε στην Επιτροπή σας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ε, ένας διεθνής ιστός ε, πρόθεσης αυτής της εργασίας Δηλαδή δεν έχουμε ένα πλήρες σχέδιο, αλλά έχουμε ένα και περισσότερα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις νέες εμπορικές συμφωνίες, στις αναπτυξιακές, στην αναπτυξιακή συνεργασία, στην συμπεριφορά των κυβερνήσεων και ε, δηλώσεις του ILO για τις ε, ΜΜΕ Πρόκειται λοιπόν για ένα ολοένα και πιο εύρωστο πλαίσιο και αυτό το βλέπουμε και στις εμπορικές συμφωνίες γιατί έχουμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες όπως το TTIP Άρα μπορεί κανείς να χτίσει αυτό τον ιστό διεθνούς δικαίου που θα μας δώσει τα θεμέλια έτσι ώστε όλη αυτή η εργασία να γίνει πιο εύκολη γιατί όλο ένα και περισσότερες χώρες θα σέβονται αυτό το πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένας πολυσχηδής χαρακτήρας των προσπαθειών. Ε, έχω πολλές τραυματικές εμπειρίες από τις προσπάθειες συντονισμού με την Παγκοσμία Τράπεζα, το ILO και ούτω καθεξής, αλλά, πάση περιπτώσει, αυτός ο ε, περίπλοκος χαρακτήρας και αυτός ο πολυσχεδής χαρακτήρας μας οδηγεί σε αυτά αποτελέσματα. Δεν ζητά κανένας άλλος το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που παρευρεθήκατε εδώ σε αυτή τη συζήτηση. So, liebe Kolleginnen Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, ακολουθείτε το υπαριθμό 6 της ημερησίας διατάξεως. Δηλαδή οι συνεχιζόμενες ε, διαπραγματεύσεις για το τριμερή διάλογο. Δύο τριμερείς διάλογοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ένας για την ε, γνωστή νομοθεσία κατά των βασανιστήριων εδώ εισηγείται η κυρία Σάκε, όπου εκεί φαίνεται να υπάρχει σημαντική προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών. Διεξάγονται τεχνικές συνεδριάσεις. Στις 16 δε Μαρτίου θα γίνει η επόμενη συνάντηση τριμερούς διαλόγου. Νομίζω λοιπόν ότι η εικόνα συνολικά είναι θετική. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος έχει ως θέμα τα ορυκτά συγκρούσεων με εισηγή τον κύριο Βίνκλερ. Εκεί δεν διαφαίνεται σύντομο το τέλος των διαπραγματεύσεων διεξήχθη το διάλογο στην 1η Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Υπό την ε, διεύθυνση του κυρίου Βάντερμπεργκ του Ολλανδικού Αρμόδιου Υπουργείου με παρουσία μάλιστα και της ίδιας της Επιτρόπου η οποία υπέβαλε κάποιες ενδεχόμενες συμβιβαστικέ προτάσεις. Διεξήχθη σε θετικό κλίμα συνεργασίας ότι τριμερής αυτός διάλογος, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικές θέσεις σε ορισμένους τομείς και ιδίως ό,τι αφορά την δεσμευτικότητα και την συμμετοχή επιχειρήσεων. Για την ώρα δεν έχουν οριστεί άλλες ε, ημερομηνίες για τις συναντήσεις. Εγώ τουλάχιστον κατέστησα σαφές απέναντι στο Συμβούλιο ότι αν δεν διαθέτει διαπραγματευτική εντολή δεν έχει νόημα να οριστεί από τώρα η ημερομηνία για τον επόμενο τριμερή διάλογο. Τώρα το περίφημο μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Συμβουλίου το οποίο θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μάλλον δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Στην πληροφορία που μόλις μας δώσατε, ε, ήταν έτσι τα γεγονότα. Και ό,τι νεότερο προκύψει ε, στο θέμα αυτό, θα μας το πει μάλλον το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να πάρει το μπαλάκι και να παίξει. Μπορούμε βεβαίω και εμεί κάποια στιγμή να οργανώσουμε τι εσωτερικέ μα συζητήσει, όμω η στιγμή αυτή δεν έφτασε ακόμη. Πρέπει να περιμένουμε το τι θα κάνει το Συμβούλιο, έτσι όπω έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Νομίζω, βάσει και το δικού σα του συντονισμού και όπω είπατε, να παραμένουμε στη συγκεκριμένη εντολή που έχει προψηφίσει η Ολομέλεια και εφόσον τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του Συμβουλίου απέχουν πολύ από τη θέση του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να περιμένουμε. Πριν συναντηθούμε μεταξύ μας και προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τις δικές μας διαφορές απόψεων, διότι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές ομάδες δεν ε, έχουν ακριβώς όλες την ίδια άποψη, έχουν κάπως διαφορετικούς στόχους. Νομίζω για σήμερα αυτό αρκεί, αλλά μετά την πρώτη κίνηση του Συμβουλίου μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ, όπως είπατε, το μπαλάκι είναι στο τερέν του Συμβουλίου. Όσο στις επιτροπές ΣΥΝΤΑ είχα την ευκαιρία να απευθύνω το λόγο προσκεκλημένος των Υπουργών στο Άμστερνταμ και δήλωσα ότι το Συμβούλιο είναι εκείνο που πρέπει να κινηθεί τώρα και να δώσει διαπραγματευτική εντολή στην Ολλανδική Προεδρία ώστε να μπορέσει αυτή πραγματικά γνήσια να διαπραγματευτεί μαζί μας. Αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Κατέστα επίσης σαφές ή μάλλον αντελήφθην σαφώς από την πλευρά της Ολλανδικής Προεδρίας ότι ενδιαφέρεται να προχωρήσει και να ολοκληρώσει. Είναι καλό αυτό, είναι αυτό για μας, ότι οι Ολλανδοί δηλαδή έχουν τη διάθεση να κινητοποιήσουν το Συμβουλίο. Γνωρίζετε ότι η Ολλανδική Προεδρία έχει επιλέξει το θέμα των δίκαιων και έντιμων, από το ακριβού fair δηλαδή, αλυσίδων παραγωγής. Και αυτό ε, προσπαθεί να κάνει η Ολλανδική Προεδρία. Βεβαίως όλοι εμείς καλούμεθα να παρακινήσουμε και τις δικές μας κυβερνήσεις των υπολείπων χωρών μελών να συμπράξουν. Καλώς, λοιπόν εδώ λίγη το υπαριθμόν 6. Θα διακόψω μέχρι τις 5 και θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ. Διακόπτει ο κύριος Γκάσπαρη.